very happy to see a lot of guests. I hope you all managed to... ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε εδώ πολύ κόσμο. Ξέρω ότι ίσως δεν είναι καλό ότι είστε όλοι μαζεμένοι εκεί συνοστισμένοι στο πίσω μέρος της αίθουσας ενώ υπάρχουν κενά καθίσματα μπροστά αλλά τι να κάνουμε αυτοί είναι οι κανόνες. Καθίστε πάντως στα πίσω έδρανα, ακόμη και αν λένε, συμβούλιο, κομισιόν, νομική υπηρεσία κτλ. Τέλος πάντων, αυτό μην το επαναλάβετε, off the record ήτανε. Okay, thank you very much for being here. My name is Judith Sargentini. Λέγομαι Judith Sargentini. Είμαι ευρωβουλευτήνα στην ομάδα των Πρασίνων και πραγματικά να πω και κάτι τι άλλο αν ε, πράγματι δεν υπάρχουν θέσεις και οι θέσεις χρειάζονται για να μπορείτε να να ε, η είναι πολύ σημαντική για να μπορείτε να ακούτε τη διερμηνία γιατί υπάρχουν πολλές γλώσσες λοιπόν υπάρχει και μια αίθουσα ακρόασης στον τρίτο όροφο από πάνω ε, στην αίθουσα 3G3 στον τρίτο όροφο αν ε, δεν υπάρχει θέση εδώ μπορείτε να πάτε στην αίθουσα αυτή λοιπόν τώρα έχουμε καθυστερήσει λιγάκι um, so θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω αμέσως με, κάνοντας μια εισαγωγή έχουμε δύο πάνελ και μία παρουσίαση από τον Επίτροπο Ντεχούχτ για την ε, πρωτοβουλία που αναλαμβάνει σχετικά με ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Λοιπόν, να σας πω ότι φέτος ήταν, η χρονιά ήταν πολύ καλή για το, σε σχέση με το θέμα της διαφάνειας και της αξιοπιστίας η σχετική οδηγία η οποία αντιστοιχεί με τον Αμερικάνικο νόμο Dodd Frank ε, πέρασε αυτή τη στιγμή συζητούμε την υποβολή εκθέσεων ε, για θέματα μη χρηματοπιστωτικά, non-financial ε, reporting. Θα ακούσετε από τον κύριο Ντεγκούχτ πολλά πράγματα για τα ορυκτά όλες μες περιοχές. Θα ακούσετε και ε, άλλους εκπροσώπους από το φλέχτ παραδείγματος χάρη γιατί, που σχετίζεται με τα δάση. Θα ακούσετε και ε, πολλά πράγματα από διάφορες περιοχές εγώ είχα ασχοληθεί λίγο με τη, διαδικασία Κίμπερλι για τα α, διαβάντια, διαμάντα από εμπόλεμες περιοχές, τα περίφημα conflict diamonds και θα τα πούμε όλα αυτά για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να προχωρήσουμε και να προτείνουμε νομοθετικές ε, πράξεις ε, αλλαγές στην νομοθεσία και στη, σε αυτό που συμβαίνουν παραδοσιακά θα μου πείτε πως μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά όχι δεν μπορούν να αλλάξουν αλλά μπορούμε να κάνουμε τις προτάσεις μας για να προχωρήσουμε πιο κοντά στη βιώσιμη ε, ανάπτυξη αν θέλετε αυτού του κλάδου εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μάθω όπως και εσείς. Κανείς δεν βρίσκεται εδώ για να μας παρουσιάσει απλώς τις απόψεις του. Όλοι πρέπει να μάθουμε και γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκονται πολλά άτομα στην αίθουσα. Και πραγματικά ε, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε ε, αμέσως γιατί καθυστερήσαμε δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας πρέπει να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα ε, αρχίζω κατευθείαν με το πρώτο πάνελ που έχει τίτλο ε, τις εξοριστικές βιομηχανίες και το ρόλο τους στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη, προκλήσεις και ευκαιρίες που υπάρχουν. Ο, την ο κύριος Τέτε Χορμέκου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Γκάνα θα μας κάνει την πρώτη παρουσίαση. Κύριε Χορμέκου καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες έστω και όχι με τη φυσική σας παρουσία. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί δεν μπορούσατε να είστε εδώ αλλά χαιρόμαστε που είστε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Κάνα για να μας μιλήσετε. Ο κύριος Χορμέκου είναι επικεφαλής του προγράμματος για το Διεθνές Εμπόριο και θέματα οικονομικής πολιτικής στη Γραμματεία για την Αφρική του ε, Δικτύου ε, του τρίτου κόσμου για την Αφρική και έχετε ασχοληθεί με οικονομικά βέβαια επενδύσει ε, και θέμα, ασχολείστε με θέματα εμπορίου από το 96 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ο τίτλος σας το τίτλος της ομιλίας σας είναι γιατί η ο ορυκτός πλούτος της Αφρικής δεν κατάφερε να συνδράμει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Υπήρου. Έχετε γύρω στα 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Θα σας παρακολουθούμε βεβαίως, αλλά δεν πρόκειται να σας διακόψουμε από εδώ. Φροντίστε να τηρήσετε τα 10 λεπτά και μετά την ομιλία ε, μετά από εσά θα μιλήσουν άλλοι δύο ομιλητές και μετά θα υπάρξει ένας κύκλος ερωταπαντήσεων. Λοιπόν, ο λόγος εσάς κύριε Ορμακού. I can't hear you now, so maybe somebody can help me. Δεν ξέρω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 Okay. So I was going Λοιπόν, θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας από την Κάνα, στις Βρυξέλλες. Ε, δεν έχω και πολύ χρόνο, γι' αυτό θα μπω κατευθείαν στο θέμα μου. Όλοι ξέρουμε ότι το θέμα που συζητούμε είναι που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Ο ήχος όμως δεν είναι καλός, γι' αυτό οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Growth, dramatic growth rates that have taken place in Africa driven by the mineral exploration and mineral exports. So it is very justifiable to ask ourselves why is it that in the face of this dramatic boom in mineral production and exportation we still have massive poverty, joblessness,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 should remove themselves from direct intervention in the mining sector. Now, and they also have to, you know, prevent. I I have to ask you to conclude. I've been giving. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, διότι θα σε έδωσα κάποια πρόσθετα λεπτά ομιλία, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα που πραγματεύεστε, αλλά παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Conclude by saying this. So unfortunately what we have is that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 πολύ διδακτικό το συμπέρασμα που αντλήσατε. Ε, μιλάτε για τη χαμηλή φορολογία των εξορρυκτικών βιομηχανιών στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και μιλήσατε και για τους εξαγωγικούς δασμούς ε, των πρώτων υλών που έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, εξάγονται λοιπόν οι πρώτες ύλες από τις χώρες σε υπερβολικά χαμηλή τιμή. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι υποφελή συναλλαγή για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είπατε βέβαια και πολλά περισσότερο όχι μόνο αυτά, αλλά ε, αυτό τουλάχιστον με ε, ε, σημάδεψε. Το, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε και τους υπόλοιπους ομιλητέ μας και θα επανέλθουμε σε εσά. μόλις ολοκληρώσουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σαρμέκου. Τώρα ο επόμενος ομιλητής, ένα λεπτάκι να βρω τα χαρτιά μου και πάλι, είναι ο Σέρχιο Άντρες Κορονάντο Ντελγάντο. ο οποίος είναι ειδικό στο συνταγματικό δίκαιο. Επίσης έχει μάστερ στην ανάπτυξη της υπέτρου και τώρα είναι συντονιστής ε, για τα δικαιώματα γης στο ΣΥΝΕΠ ε, που είναι ένα κέντρο έρευνας για την δημοκρατία και την... Ε, λαϊκή εκπαίδευση ε, έχει ασχοληθεί με την πολιτική, τις πολιτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ άλλων. Θα μας μιλήσει για τις εξορρυκτικές ε, βιομηχανίες στη Λατινική Αμερική. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι το προσέξατε εξάλλου ότι δεν μεταφράστηκε η ομιλία από τα αγγλικά. Αυτό οφείλεται στην απόσταση που μας χωρίζει και τον ε, μη ικανοποιητικό ήχο στην τηλεδιάσκεψη. Όλες οι υπόλοιπες ομιλίες θα μεταφραστούν ως συνήθως. Ε, Σέργιο, σε ακούμε για 10 λεπτά. Μπορείς να διαλέξεις όποια γλώσσα θέλεις, αλλά να ανάψεις το μικρόφωνο. Yes. Okay. Muchas gracias por Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με προσκάλεσε έτσι ώστε ε, να ε, συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, αναφέρεται και στις σκέψεις και τα συμπεράσματα της Κολομβιανής Πλατφόρμας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημοκρατίας και Αναπτύξεως που ασχολείται με τα ανθρώπινα και πολιτιστικά και αναπτυξιακά δικαιώματα στην Κολομβία τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει λοιπόν τα τελευταία χρόνια για, για την εξαγωγική βιομηχανία τις εξορυκτικές συγγνώμη, δραστηριότητες. Ε, η ε, απεικιοκρατική ιστορία της Λατινικής Αμερικής ε, έχει αποκαλύψει μεγάλες δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με την εξόριξη. Στην Κολομβία η παρούσα κοινωνική αντίδραση όσον αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες αναπτύσσεται βασιζόμενη βασιζόμενη σε ακριβώς αυτήν την ιστορία. Ε, πρέπει να σας πούμε ότι μέσα σε μία δεκαετία ε, ε, η εξόριξη άνθρακα από 38 εκατομμύρια 242.000 τόνους τον χρόνο έχει περάσει στα 74.350.000 εκατομμύρια τόνους το 2010. Ε, επίσης έχει αυξηθεί ε, με τρομακτικό τρόπο η επιφάνεια, ε, η εκμεταλλευόμενη επιφάνεια. Έχουμε περάσει από 1,1 εκατομμύρια εκτάρια το 2002 σε 8,4 εκατομμύρια εκτάρια το έτος 2009 οι κοινωνικές εντάσεις οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία ε, εξορυκτικών βιομηχανιών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ανάμεσα στον Ιανουάριο του 2001 και τον Δεκέμβριο του 2011 έχουν καταγραφεί 274 διαφορετικές μορφές κοινωνικού αγώνα που σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου, χρυσού και άνθρακα. Αυτές ε, οι κοινωνικές ε, μάχες, αυτοί οι κοινωνικοί αγώνες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια μιας διαδικασίας και ενός σεναρίου καταπολέμησης οποιασδήποτε ε, αντίδρασης και διαμαρτυρίας. Ε, μεγάλης κλίμακας εξορυκτική δραστηριότητα στην ε, Κολομβία δεν βοήθησε την υπέρβαση ε, της ένδυας στην Κολομβία και δεν επέτρεψε την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Αντιθέτως πρέπει να πούμε ότι η ο λόγος ανάπτυξης της ε, εξόριξης ε, του άνθρακα είναι αντίθετα ανάλογος ε, με τον βαθμό κάλυψης των βασικών και θεμελιωδών αναγκών του πληθυσμού. Αυτή η κατάσταση βεβαίως έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά και την εσωτερική οικονομία της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι έχουν δοθεί πάρα πολλές παραχωρήσεις προχωρήσει στην εξωτερική βιομηχανία ε, με μειώσεις ε, των ε, φόρων που πρέπει να πληρώσουν κτλ και πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την αγροτική οικονομία και την οικονομία της υπαίθρου ε, κοινότητες της ε, υπαίθρου έχουν δει το επίπεδο ζωής τους ε, να χαμηλώνει λόγω και της μόλυνσης του εδάφους και της μείωσης της ποιότητας των υδάτων. Έχουν στραφεί λοιπόν προς τους δικαστές πλέον οι πληθυσμοί αυτοί και τα τελευταία 20 χρόνια έχουν έχουν ξεκινήσει, έχουν αρχίσει να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη. Επίσης πρέπει να πούμε ότι 3.500 οικογένειες αυτοχθόνων ζενού ε, στην περιοχή της ε, Κόρδοβα έχουν ε, ξεκινήσει συγκεκριμένες ποινικέ διαδικασίες μέσω μηνύσεων κατά της Θέρο που είναι μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται το σίδηρο και τον νικέλιο σε εκμεταλλεύσεις ιδιοκτησίας BHP Billington αγγλικού κεφαλαίου. Θα ήθελα να μιλήσω και, να συσχετήσω την δραστηριότητα της εξόριξης με τους εκτοπισμούς πληθυσμών. Ε, τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε δει σημαντικές ε, αλλαγές όσον αφορά την χωροταξία ε, και όσον αφορά και τους πληθυσμούς που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πούμε ότι οι περιοχές όπου υπάρχουν ε, ε, εξορυκτικές δραστηριότητες είναι ακριβώς οι περιοχές τις οποίες είχαμε και τα τελευταία 50 χρόνια την ε, στρατιωτική παρουσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι και διαπιστώνουμε ότι 80% των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στην Κολομβία παρουσιάζονται σε τις περιοχές με πετρελαϊκή και εξορυκτική δραστηριότητα. 87% ε, του υποχρεωτικού εκτοπισμού προέρχεται από αυτές τις κοινότητες. 78% των ε, εγκληματικών ενεργειών κατά συνδικαλιστών, 89% ε, των ε, εγκληματικών ενεργειών κατά αυτοχθόνων πληθυσμών, καθώς επίσης και 90% κατά των εχόντων αφρικανική καταγωγή. Όλα αυτά τα εγκλήματα γίνονται ακριβώς σε, αυτές, σε αυτούς τους θύλακες των ορυχείων. Τώρα, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση ανάμεσα στην εξορεκτική ε, διαδικασία ε, και την ευαισθησία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διαφόρων εθνοτικών ομάδων. Σύμφωνα με την Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κολομβίας, το σύνολο των συλλογικών εδαφών των ε, μαύρων ε, κοινοτήτων έχουν ε, αναγνωριστεί ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραχωρούν στο κράτος τις, τα δικαιώματά τους όσον αφορά την εξορρυκτική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ μικρή η πληροφόρηση που έχουν οι πληθυσμοί αυτοί και δεν λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα των ιδίων πληθυσμών στην ε, τελευταία ε, έκθεσή του ε, η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τελευταία έκθεση για την Κολομβία καταγράφει ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη διαδικασία έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση και έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθότερες πρακτικές. Σε ε, μεγάλο βαθμό πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ε, οι εξορρυκτικές ε, διαδικασίες είναι σημαντικές για το γενικό καλό και για το κοινωνικό γενικό όφελος. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις μεγάλων προβλημάτων καθώς επίσης και μεγάλων διαφωνιών όσον αφορά τις εξορρυκτικές ε, διαδικασίες με την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό στην ουσία ε, καταργούνται πάρα πολύ μεγάλες επιφάνειες και αφαιρούνται από την ε, γεωργία καθώς επίσης και από την συντήρηση του περιβάλλοντος και επομένως δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται διαρκώς αποφάσεις οι οποίες θα είναι υπέρ της εξορεκτικής διαδικασίας και προς ζημίαν όλων των υπολείπων δραστηριοτήτων. Πρέπει να πούμε ότι στην έκθεση που ανέφερα προηγουμένως της εισαγγελίας της Δημοκρατίας ε, κρούεται ο κόδωνος του κινδύνου όσον αφορά ε, το κόστος το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ βαρύ ε, σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουν δοθεί και τις άδειες για εξόριξη. Διότι αυτές οι άδειες οι οποίες μεγαλώνουν όλο και περισσότερο τελικά αποβαίνουν επιζήμιες για την τοπική οικονομία για την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα του νερού κτλ ε, την ε, βιοπικιλότητα κτλ. Ε, σύμφωνα με το, την έκθεση αυτή, ε, οι εξορυκτικές δραστηριότητες ε, είτε γίνονται σε στοές, είτε γίνονται επιφανειακά, είτε είναι νόμιμες, είτε είναι παράνομες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονται κατά των οικοσυστημάτων και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, τα δάση, την γεωργία κτλ. αλλά και μέσω της σε ποιότητα του αέρα δημιουργούν προβλήματα στην ίδια την ανθρώπινη ε, ζωή. Ε, γι' αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις. Ε, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν, να γίνουν προτάσεις βάσει και των προτάσεων που, έκανε, που έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη στην δικιά τους έκθεση έτσι ώστε να φτάσουν και ενώπιον της δικαιοσύνης πραγματικά περιπτώσεις κατάφορες παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παραβιάσεις σχετιζόμενες με την εξορεκτική διαδικασία ε, θα πρέπει οι υποθέσεις ε, αυτές να λαμβάνονται υπόψη και να συζητούνται στα εθνικά δικαστήρια. Επίσης, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει ε, ε, και να υποχρεώσει τις ε, εξορρυκτικές βιομηχανίες, τις εταιρείε δηλαδή οι οποίες ασχολούνται με την εξορρυκτική βιομηχανία, να δημοσιεύουν τις τακτικά εκθέσεις όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν στην Κολομβία. Ε, η Κολομβία μάλλον είναι μια χώρα ε, η οποία υποφέρει από την στρατιωτική ε, παρουσία και τις στρατιωτικές διενέξεις και επομένως δεν είναι δυνατόν να ζημιώνεται ακόμα περισσότερο και από οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε ε, να αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος μιας ε, πρωτοβουλίας ε, η οποία ακριβώς θα είχε στόχο την σωστή αντιμετώπιση του θέματος. Θέλουμε η εξόριξη να αποβαίνει τελικά οικονομικά ωφέλιμη για τους ντόπιου πληθυσμούς και να γίνει με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι αρχές της αηφόρου ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Sergio. And I... Πολύ σας ευχαριστούμε και αυτό που πρόσεξα στο τέλος είναι όλοι γίνεστε πολύ συγκεκριμένοι στα συμπεράσματά σας. To get access, getting access. Αλλά επιμείνατε για το θέμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη όχι μόνο στη χώρα όπου γίνεται η εξόριξη, αλλά και στη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της εξορρυκτικής επιχείρησης. For Και Μας μιλήσατε για το, τη ΣΕΛ στη ΣΥΠΑ και τη Royal Dutch Shell ε, στην Ολλανδία. Δεν είχαμε την έκβαση που όλοι επιθυμούμε, αλλά Κατανοούμε ότι είναι απαραίτητες οι αξιολογήσεις και οι κοινωνικές, ε, κοινωνικού χαρακτήρα δημοσκοπήσεις. Ας συνεχίσουμε τώρα με τον ε, Σάσκια Οζιγκα που εργάζεται για το ΦΕΡΝ. Να μου εξηγήσετε και τι είναι το ΦΕΡΝ, γιατί δεν το βρήκα. Ασχολείστε όμως με παγκόσμια ζητήματα δασοκομείας και γενικότερα ευρωπαϊκά ζητήματα. Βιολογία έχετε σπουδάσει στην Ουτρέχτη και έχετε ασχοληθεί και με περιβαλλοντικά ζητήματα και φοιτήσει σε διάφορα πανεπιστήμια. θα μας μιλήσετε για τις ε, ε, λήψεις των VPAs, ε, δηλαδή των Συμφωνιών Θελούσιας Εταιρικής Σχέσης. Σα, σας ακούμε. Τι σημαίνει φέρν, τίποτα. Μας άρεσε απλώς και Ε, και μας άρεσε γιατί σημαίνει φτέρι, αλλά δεν είναι ακρονίμιο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας μιλήσω για τις ε, ελλείψεις ε, των ε, συμφωνιών αυτών στον τομέα της εξορρυκτικής βιομηχανίας. Θα ήθελα να κάνω τέσσερις βασικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα όμως να διευρύνουμε κατά τη συζήτηση και να μην ασχοληθώ μόνο με τα VPAs. Πρώτη παρατήρηση είναι η λογική συνέχεια των δύο προηγουμένων παρεμβάσεων. Δηλώνω λοιπόν το εξή ότι για να προάγουμε την ανάπτυξη μέσα από υπεύθυνε εταιρικέ πρακτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει πώ θα ορίζει και θα μετρήσει την ε, ανάπτυξη, το, η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι το σωστό το ε, μέτρο και αυτές οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης δεν είναι το σωστό εργαλείο. Για Βλέπω ότι πλησιάζουμε το 2014 και πολύ λίγα ακόμη συζητούνται εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και γενικότερα στο Δημόσιο Διάλογο για την επίπτωση αυτών των VPAs επί της ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι επίσης ότι δημοσιεύθηκε χθε ένα άρθρο στους Financial Times και ο Επίτροπος Ανάπτυξης σωστά είπε ότι λόγω της ελλείψεως θέσεων απασχόλησης στην ποσαχάρη Αφρική έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αστάθεια, σειράξεις, ε, μαζικές ε, μεταναστευτικές ε, ροές, ε, αλλά το βασικό που είπε στο άρθρο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια, ένα θετικό αναπτυξιακό θεματολόγιο. Μας εξήγησαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές ότι αν ε, η οικονομική μεγέθυνση δεν μας οδηγεί απαραίτητα σε ανάπτυξη, διότι δεν αφορά όλους και άρα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως μέτρο για τη βιομηχανοποίηση της χώρας. Ναι, έχουμε διάφορα δίκτυα που έχουν εξαγάγει μελέτες για την Αφρική και μας δείχνουν ναι, ότι είναι ανθή η οικονομία στην Αφρική, το διαβάζεται παντού, όμως δεν υπάρχει βιομηχανοποίηση και ε, πέφτει ο αριθμός των μεταποιημένων αγαθών. Οπότε η οικονομική μεγέθυνση τι σημαίνει, ότι όσο το δυνατόν γρηγορότερο γίνεται να απομυζήσουμε τη χώρα και στη συνέχεια να φύγουμε. Η δεύτερη δήλωση, γιατί δεν έχουμε και χρόνο και ε, πρέπει να μιλάω γρήγορα, για να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσα των εξορρυκτικών βιομηχανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει τι συστάσει ε, τη αναθεώρηση για την εξορρυκτική βιομηχανία. Η Παγκόσμια Τράπεζα ζήτησε αυτή τη μελέτη το 2001 για να θεωρηθεί ω εφαλτήριο και να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο αυτέ οι συστάσει. Νομίζω ότι όλοι ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα το 2003. Θα γνωρίζουν αυτά που θα πω. Τέλο σα διαβάζω δύο-τρει προτάσει από την έκθεση του πάνελ. Η έκθεση κάνει τέσσερι συστάσει σε σχέση με το πώ μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και την εξαιρετική βιομηχανία αφενό και το κράτο ε, ε, αφετέρου. Ε, είναι φτωχή η δημόσια διακυβέρνηση στον τομέα τη εξαιρετική βιομηχανία, και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Στη συνέχεια πρέπει να ενισχυθούν οι παρεμβάσει Παγκόσμια Τράπεζα στον τομέα αυτό και τρίτον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση θα δείτε ότι εστιάζεται γύρω από την κεντρική ιδέα ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να υποστηρίζει την εξαιρετική βιομηχανία μόνο στο μέτρο που συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο μήνυμα τη έκθεση. Πολλά μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία και από τι συστάσει ε, τη αποτίμηση ε, που έγινε. Όπω είπε και ο προηγούμενο ομιλητή, ε, υφίσταται πάρα πολλά προβλήματα. VPA, συμφωνίε εθελοντική εταιρική σχέση. Μου ζητήσατε να σα μιλήσω για τι ελλείψει των VPA. Ναι, αλλά είναι και το πλέον ρηξικέλευτο εργαλείο που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να δώσει ε, μία απάντηση, να αντιδράσει σε σχέση με το στόχο των ε, καλών εταιρικών πρακτικών. Όντω, ε, είναι εστιασμένε γύρω από τη λογοδοσία και τη διαφάνεια οι VPAs. Αλλά να σα ρωτήσω, ξέρει κανεί εδώ μέσα τι είναι μία VPA. Εάν ξέρετε, μπορείτε να σηκώσετε το χέρι, παρακαλώ, αν γνωρίζετε τι σημαίνει VPA. Η μισή περίπου. ούτε καν, έτσι. Πρωτό να σας πω τίποτα για τις ελλείψεις, μάλλον να ορίσουμε τις VPS, να ξέρουμε και τι είναι. Ε, voluntary Partnership Agreement ε, είναι μια, είναι μια δεσμευτική εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί με έξι χώρε η Ευρωπαϊκή Ένωση προ το παρόν και τώρα <coughs> διαπραγματεύεται με άλλε 7 και άλλε 10 είναι σε προ-διαπραγματευτική φάση. Ο στόχο είναι να ελέγξουμε την παράνομη υλοτομία σε αυτέ τι χώρε και τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει αυτών των χωρών θα καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να ορίσουν τι εστί νόμιμο και τι εστί έκνομο, στη συνέχεια ένα σύστημα ώστε να ανοιχνεύουν μαζεύουμε το ξύλο από την παράνομη υλοτομία σε όλη την τροφοδοτική αλυσίδα για να ε, εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο νόμιμο σε εισαγωγικά ξύλο και στη συνέχεια μια εποπτική διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά συναπαρτίζουν την Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Ο στόχο όμω του VPA, η βάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ότι ε, πρέπει να ενισχύσει την, το ρόλο των κυβερνήσεων, να ενισχύσει ε, τα δικαιώματα μίσθωση του εγχωρίου πληθυσμού να ενισχυθεί η διαφάνεια και όλα αυτά τα, συ... τα σχετικά. Ναι, πέρα από το σύστημα ανείχνευσης και ελέγχου, και αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας, ε, τι έχει γίνει όμως. Ενισχύεται η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις της και μετέχουν στις διαπραγματεύσεις ε, αυτών των συμφωνιών, άρα είναι μάλλον επαναστατικής φύσης αυτό το εργαλείο και ε, ήθελα να πω βεβαίως ότι αυτό πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο για άλλου είδους εμπορικές συμφωνίες που τώρα διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι EPA, παραδείγματο χάρη, και άλλου είδους συμφωνίες δεν διαπραγματεύονται, ε, χωρί, δεν ε, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση χωρίς ε, αποκλεισμούς και αυτό θα γυρίσει μπούμερανγκ εν τέλει, κατά τη γνώμη μας. Θα ήθελα να σας πω και για αυτό αυτό το θέμα, για τις ελλείψεις λοιπόν ε, και τις αδυναμίες του VPA. Ε, είναι ξεκάθαρο αν δείτε τι συμβαίνει στη Λιβύρια, στο Καμερούν. Ε, ο τομέα τη υλοτομία είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι χώρε και τα τελευταία χρόνια σε σημασία, ενώ ο γεωργικό τομέα έχει αυξανόμενη σημασία. Αν δείτε τις εισαγωγές προς Ευρωπαϊκή Ένωση. At the moment come from conversions from agricultural, uh, agricultural concessions rather than from forest concessions. Μεγαλύτερα νούμερα τα βλέπουμε όχι από παραχωρήσεις γης από, αλλά από εταιρείε που δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό είναι μια πρώτη αδυναμία γιατί δεν υπάρχει μετοχή της ε, τοπικής κοινωνίας. Δεύτερον, οι VPAs συνδέονται με την κείμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση για τα ξύλα. Ξέρετε, ποιο, ποιοι ξέρουν τι είναι, ποια είναι η νομοθεσία. Α, πολύ περισσότεροι. Λοιπόν, η νομοθεσία Τίμερ ε, καθιστά πολύ δυσκολότερο το να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο παράνομα τέτοια ξύλα. Ε, το πρόβλημα με την UTR είναι ότι δεν εφαρμόζεται ακόμη με σε ικανοποιητικό βαθμό σε επίπεδο ε, κράτους μέλους και αν δεν βελτιωθεί η υλοποίηση τότε ε, θα μειωθούν και οι δυνατότητες που έχουν κάποιες νότιες χώρες να διαπραγματευτούν τέτοιου είδους συμφωνίες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σταματήσω εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ Σάσκια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί τις ε, συμφωνίες EPAs. Μία ε, για την Ανατολική Αφρική και μια άλλη για, τη Καμερούν, για το Καμερούν και εγώ προ, πρότεινα να πούμε και όχι μάλιστα η, Διεθνή, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όμως δεν συμφώνησε μαζί μας ως, με την Επιτροπή Ανάπτυξης δηλαδή ε, Τώρα υπάρχει και μια EPA για την μεσημβρινή Αφρική, τεράστια η συζήτηση σχετικά. Λοιπόν, τώρα σας πρότεινα χρόνο για ερωταπαντήσεις. Σας είπα ότι θα μιλήσει και ο Επίτροπος Δεχούχτ Εγώ λέω να μιλήσει πρώτα ο Επίτροπος Δεχούχτ και μετά να προχωρήσουμε στο κομμάτι των ερωταπαντήσεων. Επίτροπε Ντεχούχτ, ελάτε εδώ. Υπάρχει μια θέση δίπλα από το Σέργιο. Um, uh, Ο Επίτροπος Τεχούχτ θα μιλήσει για την πρωτοβουλία του σχετικά με ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Ορυκτά και μεταλλεύματα από εμπόλεμες περιοχές. Good morning. Uh, Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, συμμετέχοντες σε αυτήν την συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνεται να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Είμαι πάντα ευτυχής όταν ε, μπορώ να μιλήσω ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θυμούνται φαντάζονται, φαντάζομαι και τα ε, μέλη της ε, Επιτροπής ε, Ανάπτυξης ε, ότι 14 χρόνια ήμουν και εγώ ο ίδιος βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, το θέμα σήμερα είναι η συζήτηση αυτή για την σχέση ανάμεσα στον ρόλο που μπορούν να παίξουν ε, η εξόριξη των πρώτων υλών, να μπορεί να παίξει η εξόριξη των πρώτων υλών ε, στην ε, ανάπτυξη ε, βεβαίως αυτή η, αυτό, αυτό το είδος εμπορίου θα πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για οποιαδήποτε αναπτυσσόμενη χώρα ε, ε, να δίνει τη δυνατότητα για εισρωή χρημάτων στην οικονομία, να δημιουργεί ανάπτυξη, ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασίας ε, και μέσω των φορολογικών εσόδων χρηματοδότηση και ενίσχυση διαφόρων τομέων όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση κτλ. Βεβαίω το θέμα, όπως γνωρίζετε, είναι να μην πέσει κανεί σε παγίδες ε, ε, ε, οι οποίες τελικά να δίνουν χώρο για, την, για διαφθορά και για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο τελικά δεν θα ευνοήσει τι σωστές οικονομικές διαδικασίες. Ένα, μία από τις πιο σοβαρές παγίδες είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το, κυρίως σε εμπόλεμες περιοχές. Έχουμε δει ε, φαινόμενα περίεργα παλιότερα με τα διαμάντια και τώρα με το χρυσό και με άλλου είδους ε, ε, τιτάνιο και άλλα ορυκτά. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κόστους, του ανθρώπινου κόστους πρέπει να είναι υποχρέωση συνδεδεμένη με όλα τα προϊόντα ε, που προέρχονται από τις χώρες αυτές ε, και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση ε, λόγω της ενιαίας αγοράς που είναι μία βεβαίως από τις κυριότερες τελικές, κυριότερους τελικούς προορισμούς για αυτές τις πρώτες ύλες μπορούμε να επηρεάσουμε την ε, κατάσταση. Η διεθνής ε, κοινότητα και ε, βεβαίως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΣΑΑ, τη G8, τα Ηνωμένα Έθνη, τα, οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να ξεκινήσουν την δράση. Και εμείς βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρώπη, θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε. Ήδη ε, τώρα μπορώ να σας πω ότι λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες ε, επιλογές, επομένως δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την τελική επιλογή, γιατί το Κολέγιο των Επιτρόπων δεν έχει πάρει ακόμα σχετική απόφαση. Όμως μπορεί να είμαι πάρα πολύ σαφής λέγοντας ότι οτιδήποτε κάνουμε ε, θα οδηγείται από τρεις άξονες. Αποτελεσματικότητα, μείωση των ε, παράπλευρων ε, αποτελεσμάτων και μεγάλος συντονισμός. Πρώτα απ' όλα η αποτελεσματικότητα, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα. Η πρόκληση εδώ είναι η περιπλοκότητα. Σε αυτή την περίπτωση η περιπλοκότητα της ε, αλυσίδας ε, που ε, συνδέει τις, τα ορυχεία κύβου στο Κονγκό στην, στον εμπορικό δρόμο των Βρυξελών, τη Ρινεύ. Έχουμε δει από κοντά το θέμα αυτής ε, της ε, αλυσίδας ε, και είδαμε ότι έχει μειωθεί η περιπλοκότητα Όσο δηλαδή πιο κοντά στην πηγή βρίσκεται κανείς και μπορεί να την ελέγξει, τόσο λιγότερη περιπλοκότητα παρουσιάζεται, τόσο περισσότερο μπορεί να ελεγχθεί το προϊόν. Ε, είναι γεγονός ότι ε, η, η, τελική φάση της ε, αλυσίδας που είναι η τήξη των μετάλλων είναι αυτή η οποία μπορεί να δημιουργήσει τα περισσότερα, να δώσει τα περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να αξιολογήσουμε το πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με μια πιο σφαιρική προσέγγιση ε, στην αλυσίδα ε, προμήθειας, αλλά δεν μπορώ να είμαι περισσότερο σαφής και ακριβής. Επίσης προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ε, έτσι ώστε οι πληροφορίες ε, τις οποίες ε, συλλέγουμε να δοθούν σε, όλα, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Τα μεταλλεύματα τα οποία προέρχονται από περιοχές που βρίσκονται σε διένεξη δεν είναι βεβαίως ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται μονάχα με την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Έχουμε και άλλα παραδείγματα όπως ας πούμε τους ΦΑΡΚ στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα και τις ε, περιοχές ε, όπου δρούν οι αντάρτες ε, αυτές. Ε, έχουμε εκθέσεις ε, οι οποίες ε, μας δείχνουν ότι και το χρυσό και το ταντάλιο και το κολτάνιο εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τις εκστρατείες των ομάδων και για την παραγωγή κοκαίνης στις περιοχές αυτές. Συγγνώμη, από τη στιγμή που η διακίνηση της κοκαίνης έχει γίνει πιο δύσκολη για τις περιοχές αυτές το Ινστιτούτο Χαϊδελβέργη εκτιμά ότι 20% ε, των ε, ε, συνολικών διενέξεων σχετίζεται με τις πρώτες ύλες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, βεβαίως ε, ε, αυτό που καταλαβαίνουμε επίσης είναι ότι τα παράπλευρα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι ίσως πιο δύσκολο να τα καταπολεμήσει κανείς. Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτές τις περιοχές είναι ίσως το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους εντόπιους πληθυσμούς. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν διασφαλίσεις όσον αφορά το, το θέμα αυτό ε, και ότι εν πάση περιπτώσει ε, θα δημιουργηθεί ε, και τοπική αγορά αλλά και ασφάλεια προμήθειας. Η ασφάλεια προμήθειας όσον αφορά τις πρώτες ύλες είναι ουσιώδους σημασίας. Και εγώ, σαν Επίτροπος Εμπορίου, βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσω και να ενδυναμώσω την ευρωπαϊκή οικονομία κατά αυτή την έννοια το Λέω αυτό γνωρίζοντας βεβαίως ότι ενδεχομένως μερικοί μεταξύ ημών βλέπουν το θέμα αυτό ως λιγότερο σημαντικό. Μπορώ να τους καταλάβω, πάντως πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επιλέξουμε αυτήν την οδό. Το τρίτο μας μέλημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να είμαστε βέβαιοι ότι η πρότασή μας ε, θα ε, μπορεί ε, να ενταχθεί σαφώς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης που αφορά το ίδιο θέμα. Από τη μία πλευρά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε την ευρύτερη εξωτερική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική έτσι ώστε στις περιοχές διένεξης να έχουμε πιστοποιημένα καθαρά ορυχεία, εντό αγωγικών το καθαρά. Ε, σημαντική είναι η προσπάθεια από την πλευρά της εμπορικής ε, πολιτικής, έτσι ώστε ε, πραγματικά να έχουμε μια καλή και εποφέλή προς όλους κατάσταση. Αλλά βεβαίως το εμπόριο είναι μονάχα ένα, μια μικρή ψηφίδα στην ευρύτερη, μεγαλύτερη στρατηγική, η οποία λαμβάνει υπόψη σημαντικές, βαθιές, εθνοτικές ή ιδεολογικές μισθολογικές διαφορές, ασθενή ε, κράτη, ένδια κτλ. Επομένως όλα αυτά ε, θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία και γίνονται άλλωστε σε συνεργασία και με τη στήριξη ε, της Λέδης Άστον. Γνωρίζω βεβαίως και κατανοώ ότι πολλές ευρωπαϊκές ε, εταιρείες ε, ήδη ε, θέτουν σε αυτούς πάρα πολύ ψηλά πρότυπα για τους ίδιους αλλά και για τους συνεργάτες τους βάζοντας ένα θεματολόγιο το οποίο ακριβώς εστιάζεται στην ευθύνη για την υπευθυνότητα. Αλλά βεβαίως είναι και αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν λαμβάνονται ε, υπόψη ε, ή, ε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και εκθέσεις με συγκεκριμένες απαιτήσει προς τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείε, όπως είναι, ας πούμε, τα στοιχεία τα οποία και τα, αυτά που καταγράφονται στο Dot FRAC Section 1502 θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου ότι θα πρέπει να ε, αναγνωριστούν και να ενθαρρυνθούν όλες ε, οι ε, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να είναι κοινωνικά υπεύθυνες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε και έναν κατάλογο εταιριών οι οποίες λειτουργούν σωστά. Το ζήτημα, αξιότιμα μέλη, είναι ε, ότι υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις και πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την ενσωματωμένη παγκόσμια οικονομία. Ε, το εμπόριο έχει βεβαίως φέρει ανάπτυξη και ευημερία σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου ε, και η Ευρώπη φυσικά ε, αλλά και τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων και των αναδυόμενων χωρών έχουν βελτιώσει τα πρότυπα ζωής τους. Αλλά την ίδια στιγμή το εμπόριο φέρνει τους καταναλωτές της Ευρώπης σε άμεση επαφή με από άλλε ε, χώρε του κόσμου. Επομένως, ε, η σταθερή πρόκληση της ε, εμπορική πολιτική είναι πώς τα ωφέλη να μεγιστοποιηθούν, ενώ θα δημιουργούνται συστήματα έτσι ώστε τα αρνητικά, οι αρνητικές επιπτώσεις να μετριάζονται. Ε, με τον ε, τρόπο αυτό προσπαθεί να έχει επιτυχεί η εμπορική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθώντας δηλαδή να ε, μην υπάρχουν χρήματα. Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες μας έχουν νόημα εάν όμως καλύπτονται οι ανησυχίες τις οποίες παρουσίασαν νωρίτερα και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας μέχρι τα τέλη του έτους και προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία με την Επιτροπή ΔΕΒΕ και ελπίζω το 2014 να τα ξαναπούμε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Σα ευχαριστούμε Επίτροπε Ντεχούχτο. Should... Και θα έπρεπε πριν να αρχίσετε να είχα πει ότι εμείς μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία σας εδώ ο κύριος Πίλμπαξ και η Επιτροπος Γιώργεβα ήρθε στην Επιτροπή μας αλλά πιστεύω δεν λέμε δηλαδή ότι δεν έχουμε επιτρόπους αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εσείς εδώ μπορείτε να απαντήσετε μια-δυο ερωτήσεις εμείς θα ρωτήσουμε, εσείς θα απαντήσετε. Λοιπόν, θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για ε, ε, για την ε, ε τα ορυκτά ζώνες το να δουλέψει κανείς με αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να ε, ε, επιτευθεί πιο πριν μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης διότι θέλουμε ευρωπαϊκές εταιρείες να περνάνε τη διαδικασία της due diligence δύο φορές. Λοιπόν, και από εκεί δεύτερη ερώτηση. Κολομβία και τα λοιπά τα ακούσαμε. Αλλά έχετε άλλες χώρες κατά νουν ε, όταν λέτε ε, ρηκτά από εμπόλεμες ζώνες. νόησα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που κάναμε ε, τον Ιούνιο εμείς εδώ τη σχετική οδηγία που συζητήσαμε για, τους, ε, για τη διαφάνεια και τα λοιπά που τη συζητήσαμε και με τις ε, εταιρείε και η οποία οδηγία είναι ε, ακρογωνιαίος λίθος στην όλη ε, πολιτική του κλάδου. Εκείνο που είναι σημαντικό τώρα είναι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία αυτή. Πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες πήγαμε τον Σφόμποντα στην Γκάνα και στην Τανζανία γιατί, διότι οι χώρες αυτές είναι σχετικά σταθερές έχουν μεγάλο ορυκτό πλούτο, ιδιαίτερα πολύτιμα μέταλλα, ιδιαίτερα αέριο και διαπιστώσαμε ότι και στις δύο χώρες υπάρχει μεγάλη πολιτική βούληση για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων προς όφελον των πολιτών. Όπως ε, ακούσαμε και από την Κάνα υπάρχει φορολογικό πρόβλημα, η τοπική αυτοδίκηση ε, ε, παρεμβαίνει με κάποιο διαφορετικό διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς και υπάρχουν πολλά κέρδη και πολλά πλεονεκτήματα από αυτούς τους φυσικούς πόρους. Εμάς περιπτώσει, εδώ βλέπω εγώ δύο παίκτες, Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα πρέπει να δώσει τεχνογνωσία για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν ε, την, το know-how, δεν μπορούν να... Υπάρχει η πολιτική βούληση αλλά δεν υπάρχει τεχνογνωσία και ούτε καν για διαπραγμάτευση με τις εταιρείε, ούτε τίποτα παραπάνω άρα πρέπει να βοηθήσουμε και κάτι τι άλλο, το, θα πρέπει να πούμε στις ελίτ των χωρών αυτών πώς φανταζόμαστε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η κατάσταση. Θα πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν σωστά. Όλοι Κάσμαν, ο επόμενος ομιλητής και μετά δύο ερωτήσεις από το κοινό. Ορίστε, οι δύο πρώτοι που ζήτησαν το χέρι του. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Δεν διαφωνούμε με αυτά που είπατε. Όπως ξέρετε, εμεί εδώ πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να εμπλακούν οι κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών και οι δικές μας κυβερνήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, ανοιχτοσύνη ας πούμε διότι εάν δεν εφαρμοστούν με διαφάνεια και ανοιχτά ορισμένα πράγματα στις χώρες αυτές τότε καταραίουν οι ε, στόχοι μας τελείως και οι ελπίδες μας πρέπει να υπάρχουν κάποια κίνητρα και πρέπει να, να διατηρηθούν αυτά αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί και βιώσιμη ανάπτυξη των εταιριών. Πρόεδρος, ωραία. Σοφία Πίκολς, Global Witness. Δεύτερη ερώτηση, Ντάρακ από τους Friends of the Earth. Σοφία, ευχαριστώ, ευχαριστούμε ε, και τον Επίτροπο. Μιλώ ε, εκ μέρους μιας συμμαχίας 60 περίπου μη κυβερνητικών οργανισμών από πολλές χώρες Καναδά, Αμερική, Ζιμπάμπουε κλπ. Λοιπόν, ε, χτες εμείς ε, συμφωνήσαμε με την Κομισιόν για ένα έγγραφο θέσεις ελπίζουμε να ε, γίνουν αυτά που ζητούμε, να γίνονται οι έλεγχοι και οι εξετάσεις αν θέλετε γιατί δεν θέλουμε να προχωρούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ασχέτως ε, ποιες είναι ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομη να πω πολύ γρήγορα ποιες είναι οι τέσσερις συστάσεις που έχουμε κάνει, σας έχουμε δώσει και το έγγραφο βεβαίω. πρώτη σύσταση καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εφαρμόζεται σε όλους τους φυσικούς πόρους από όλες τις περιοχές. Δεύτερο, ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε γνωστά διεθνή εργαλεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Τρίτη σύσταση ότι θα πρέπει η προσέγγιση να βασίζεται στον κίνδυνο και στην αποτίμηση του κίνδυνου και τέταρτη σύσταση θα πρέπει να συμπληρωθούν με άλλες νομοθετικές πράξεις αυτά που ήδη ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να αποφύγουμε καταστροφή του περιβάλλοντος και να ενισχύσουμε την εξορικτική βιομηχανία σωστά στις τρίτες χώρες. Επόμενες, ε, επόμενος ομιλητής Friends of the Earth. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα να θέσω. Παρόμοιο με αυτό που έθεσε και η πρόεδρος Αργεντίνη για τη σχέση του το, ε, για τη σχέση μεταξύ της πρωτοβουλίας Κομισιόν και του νόμου Dodd Frank του Αμερικάνικου ε, ε, ερώτηση, επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση της κυρίας Αργεντίνη και ε, ρωτώ επίσης και τι επιπλέον φυσικοί πόροι πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο νόμο Dodd Frank θα μπορούσαν να περιληφθούν στη δική σας πρωτοβουλία. Um, thank you very much for. Uh, I can see here. You can. Uh, um, Thank you very much for the questions. Uh. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Επιτροπός, για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να συνδυάσω την πρώτη και την τελευταία ερώτηση, τη σχέση με το νόμο Dodd Frank. I think the weakness Νομίζω ότι η αδυναμία του Ντόρτ Φρανκ είναι συγχρόνως και η ισχύς του και το αντίθετο. Εκείνο που βλέπουμε ε, να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εφαρμογή του Ντότ Φρανκ είναι να υπάρχουν εμπάργο σε ολόκληρες περιοχές δεν επιτρέπονται εισαγωγέ από το Ανατολικό Κονγκό πλέον ας πούμε να βγει κάτι τέτοιο εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα σχετιστεί με την διαδικασία τήξης των μετάλλων μάλλον εξαγωγή μετάλλων από τήξη αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις εταιρείες στοχεύουμε το τι γίνεται πέρα από τη διαδικασία αυτή δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή από εκεί και πέρα βέβαια άμα αρχίσουμε να ε, ελέγχουμε δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις εταιρείε που είναι εκατομμύρια αλλά βεβαίως υπάρχει μια σχέση μεταξύ των δικών μας των στόχων και των στόχων του Dodd Frank Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή όλη η διαδικασία της δέουσας εποπτείας, της due diligence, θα πρέπει να, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι διαφορετική από αυτή που κάνουν οι Αμερικάνοι. Αλλά βεβαίως αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει μεταξύ της Κομισιόν και των Αμερικανών. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στις λεπτομέρειες του ε, στα πλαίσια των ε, συμφωνιών των εμπορικών αλλά ε, θα συμφωνήσετε ότι πραγματικά πρέπει να συζητηθεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε? Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε χωρίς τέτοιου είδους συζητήσεις. Και γι' αυτό που είπε η κυρία Σαρτζεντίνη ότι θα πρέπει να έχουμε πραγματική εξέταση και έλεγχο των εταιριών στα πλαίσια του due diligence έτσι όπως πρέπει να γίνει. Ο, τώρα οι Αμερικάνοι θα μας πούν ποιος έχει την υποχρέωση να την κάνει την εξέταση αυτή των εταιριών αλλά εμείς μπορούμε να πούμε τι θέλουμε να περιλαμβάνεται στη διαδικασία αλλά αυτά θα τα πούμε μέχρι το τέλος χρο... της χρονιάς. Από εκεί και πέρα για, τα, για το τι, ε, ε, τι εννοούμε όταν μιλάμε και τι περιλαμβάνουμε όταν λέμε ορυκτά ή μεταλλεύματα σε εμπόλεμες ζώνες. Ε, λαμβάνουμε υπόψη τον Βολφράδε, τον Κέλιο, τέλο πάντων όλα αυτά τα ορυκτά, αλλά υπάρχουν και άλλα βεβαίως Υπάρχουν στα, στη Μιανμάρ ε, υπάρχουν κοιτάσματα ενδιαφέροντα ε, ε, έχουμε διαμάντια στην περιοχή εκείνη αλλάζουν βέβαια οι κυβερνήσεις και οι προεδρίες, οι πρόεδροι στην περιοχή από τη μια στιγμή στην άλλη μετά έχουμε την Ιγυρία οι εξορίξεις για το γεωτρής και το πετρέλαιο είναι σημαντικές για την Ιγυρία Έχουμε μετά το Αφγανιστάνο με μεγάλη εξορρυκτική βιομηχανία. Εκεί υπάρχει και πρόκληση ασφαλείας, ε, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά ορυκτά ενδιαφέροντα. Άρα είναι, πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στο Ανατολικό Κονγκό. Ε, αυτό βέβαια δεν μας ε, τυφλώνει σε σχέση με το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς θα είμαστε πιο ευρείς στη διατύπωσή μας θα αναφερθούμε στα τέσσερα περίφημα και μετά αλλά όσον αφορά τις περιοχές θα ε, εννοείται ε, θα, είμαστε, θα είναι ευρύτερες περιοχές αυτές και από εκεί πέρα μετά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα ορυκτά ή Τώρα για την τεχνογνωσία, για το know-how. Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το know-how σαν δικαιολογία για είναι αυτό που είπατε και εσείς για τις ελίτ αυτές τις χώρες. Υπάρχουν ομάδες ανταρτών που εξορίσουν ε, ορυκτά και μεταλλεύματα. Δεν είναι μόνο ορισμένοι άλλοι που, είναι, που κάνουν εξόριξη ο κύριος Κάσμαν για αυτά που είπε. Ναι βεβαίως, κοιτάξτε είναι πολύ σημαντικό ε, αυτό που είπατε βεβαίως θα πρέπει η ITI να ελέγξει τα πράγματα και να δει τι χρήματα μπαίνουν στους προϋπολογισμούς των χωρών αλλά αυτή τη στιγμή μπει στον προπολογισμό το θέμα είναι μετά πώς χρησιμοποιείται και πώς εκτελείται ο προπολογισμό. Αυτή η πρωτοβουλία πολλές χώρες ε, συμ, ε, συνυπέγραψαν την πρωτοβουλία πολλές χώρες συνυπέγραψαν την πρωτοβουλία ITI αλλά Τέλο πάντων, ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν πάνε όλα τα χρήματα στον προπολογισμό. Αλλά από κάποιες πολυεθνικές πάνε τα χρήματα στον προϋπολογισμό διότι έχουν συναυθεί ακριβώς συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να κάνουν κάτι τέτοιο αλλά βεβαίως υπάρχουν και παραθυράκια ε, στην ITI συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν από κάποιους άλλους ομιλητές ε, ε, δεν ε, προσπαθούμε ε, αν προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να είμαστε φάνταστοι μπορεί να προτείνουμε κάτι το οποίο μπορεί να χαιρετιστεί με το με το το, το, από το κοινοβούλιο αλλά το οποίο ίσως δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα αν δεν διαβουλευτούμε με εκπροσώπους της καθημερινότητας ας πούμε με τη βάση ε, ξέρω λιγάκι τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο επανειλημμένα πήγα στην Κατάντα, στη Ρουάντε στο Ιτούρι, στο Ανατολικό Κονγκό ε, νοτιοαφρικανική δημοκρατία πέρασα και μια βραδιά στο παλάτι πώς το λένε αυτού του παράξενου του αυτοκράτορα κοιμήθηκα εκεί ναι τέλος πάντων είχα και πρόβλημα με το ρεύμα εκεί και μετά αναγκάστηκα να αρνηθώ ένα <laughs> με, μετάλλιο που θέλανε να μου δώσουν του τάγματος της ε, εθνικής αναγέννησης κάπως έτσι τέλος πάντων ε, πρέπει να, λαμβάνουμε βάλουμε υπόψη μας το τι γίνεται επί τόπου ε, το τι γίνεται στη βάση ο, ήτανε ε, το Κονγκό ήταν τέως βελγική απικία ε. ε, και πήγα επανειλημμένα εκεί. Βέβαια στο τέλος δεν μπορούσα να μπω μες στη χώρα αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη ιστορία. Ε, το θέμα πάντως για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητούμε δεν είναι πώς θα αναπτύξουμε μια θεωρία αλλά πώς πρακτικά θα εφαρμόσουμε αυτά που υπάρχουν δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα καινούριο παρόλο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αλλά το θέμα είναι να εφαρμόσουμε για να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτά που υπάρχουν μετά από διαβουλεύσεις κλπ. Πρόεδρος ε, μίλησαν εκπρόσωποι δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο και σε δύο ακόμη ενώσεις. Μπορείτε να μείνετε γι' αυτό. Ωραία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε Ντεγκούχτ, ήταν πολύ ε, ανοιχτέ και ειλικρινείς οι παρεμβάσει σα και το εκτιμούμε. Θα ήθελα να σα πω ότι τα μέλη ε, του, που εκπροσωπούμε ασχολούνται με την εξαγωγή μετάλλων, είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτό το πρόβλημα και ακολουθούν ήδη τις αρχές της εταιρικής ευθύνης, άρα μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαφάνεια στην τροφοδοτική αλυσίδα Επίσης, να ξέρετε ότι η πλειοψηφία αυτών των εταιρείων δεν έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, αλλά σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη Κίνα, Μαλαισία ε, και άρα δεν δεσμεύονται από την ίδια διαδικασία υποχρέωση επιμέλειας. Ε, τίθενται επίσης ε, σοβαρά ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Μετά την παρουσίαση του νόμου Dodd Frank, ε, η πλειοψηφία των Αμερικανικών αγορών εγκατέλειψαν ε, την αγορά και του, τις αντικατέστησαν απλώς ε, άλλες εταιρείε που δεν δεσμεύονται από αυτήν την νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε αν αυτή η νομοθετική πρόταση περιέχει ε, πρακτικές λύσεις, πώς ε, θα ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους οι εταιρείες, πώς θα μπορέσει ο κλάδος να συμμορφωθεί με αυτές τις νέες απαιτήσεις. Τα στυλ. Σας ευχαριστώ. Απευθύνω την ε, ερώτηση στον Επίτροπο Τεχούχτ. Δύο χρόνια αγωνιστήκαμε για ούτως ώστε ε, να ελέγχεται το ξύλο από το Κονγκό, από τις εμπόλεμες ζώνες. Ε, ποια μαθήματα, ποια διδάγματα έχουμε αντλήσει. Δεν πρέπει να το θέσουμε ε, στις ε, εταιρείες για να έχουμε την υποστήριξή τους ταυτόχρονα με την υποστήριξη των κρατών μελών. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει, να κάνετε έναν απολογισμό πεπραγμένο για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ε, κάνω και, και εγώ μια ειλικρινή ερώτηση. Λέει η Πρόεδρος ποιος θα τολμούσε να αρνηθεί ένα τέτοιο αίτημα. Επίτροπος Τεχούχτ. Um, first of all on the smelters. Um, ε, πρώτα απ' όλα για αυτές τις εταιρείες η τήξη του μετάλλου πρέπει να γίνεται στην ίδια την ε, χώρα. Ε, οπότε νομίζω ότι αυτό απαντά εν μέρη στο ερώτημά σας. Τώρα, για την προστιθέμενη αξία που είναι κέρδος της χώρας όπου γίνεται η εξόριξη είναι αμεληταία, το ξέρετε. στο Κατάγκα παραδείγματος χάρη. Ε, σχεδόν όλες οι εταιρείες ε, κατέβασαν ρολά, ε, διότι για διάφορους λόγους υπάρχει σύραξη και έχουν καταστραφεί εργοστάσια, μονάδες και, και στη Ζάμπια μόλις διασχίσει κανείς τα σύνορα τα ίδια. αυτά τα μεταλλεύματα πρέπει να λιώνονται στην ίδια τη χώρα αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν είναι σταθερό το καθεστώς και επικρατεί η ειρήνη, γιατί είναι θέμα κράτους δικαίου η προστασία των ε, εταιριών. Αυτό δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί. Καταλαβαίνω επίσης ότι δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε τέτοιες εταιρείες ε, παραγωγής μετάλλων. Ε, ως προς την αξία τώρα των ίδιων των μετάλλων. Ακόμη και τώρα ε, είναι πολύ μεγάλο το μερίδιο της αγοράς για τους Ευρωπαίους. Uh, Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να στοχοποιούμε τον πληθυσμό, τις εταιρείε. και ε, κατά κύριο λόγο αυτές τις εταιρείε, γιατί και η διαδικασία Kimberly δεν είναι ότι είναι πιο στεγανή, όμως παρόλα αυτά είχε θετικές επιπτώσεις σε σειράξεις όπως τη Χεραλεόνε, παραδείγματος χάρη, που σίγουρα τροφοδοτήθηκαν από τα διαμάδια, που είναι και τα ακριβότερα στην Αφρική, η ρίστο Παρόδο. Και ε, ε, σταδιακά με τη διαδικασία Κίμπερλι καταφέραμε να ελέγχουμε όλο ένα και περισσότερο τα διαμάδια. Φυσικά, να ακούσουμε ευχαρίστως ε, οποιαδήποτε πρόταση, επιχείρημα έχετε σχετικό και ούτω η αλλω συνεχιζεται η από τα ανατολικά του Κόγκο, έτσι δεν είναι. Οπότε καλωσορίζουμε οποιαδήποτε συμβολή έχετε, οποιαδήποτε μαρτυρία έχετε να καταθέσετε για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε και τον Επίτροπο Τεχούχτ που ήρθε και ήταν ε, όσο πιο ανοιχτός και ειλικρινής μπορούσε. Περιμένουμε την πρότασή σας πριν τα Χριστούγεννα, οι φωσιολογικές συνθήκες και ελπίζουμε να σας δούμε ίσως μετά τις, ε, τα Χριστούγεννα για να ξανασυζητήσουμε την πρόταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Now, recall that we had speeches, uh, uh, uh, introductions earlier and that we actually still have... Λοιπόν, ε, θα μπορούσατε να βγάλετε την παρουσίαση και να φαίνεται ο προσκεκλημένο μας από την Γκάνα και πάλι στην οθόνη. Σας παρακαλώ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις ε, για τη μη βιώσιμη εξορρυκτική δραστηριότητα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα παρακαλώ να παραμείνετε εδώ στο βήμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσετε τις ερωτήσεις που σας ενδιαφέρουν ε, προτού ε, περάσουμε ε, στις απαντήσεις και στη συνέχεια στα συμπεράσματα. Τώρα online έχουμε τον κύριο Χιορμέκο. Εδώ μαζί μας έχουμε τον κύριο Σέργιο Ανδρές και την κυρία Οζίντα. και στη συνέχεια στο δεύτερο πάνελ έχουμε την κυρία Μελό και τον κύριο Ριντόλφη. Ε, ποιος είναι εδώ για τους άλλους δύο μιλητές. Αν ήρθαν ε, εδώ όλοι για τον Επίτροπο Ντεχούχ θα μπορούσα να σας είχα ειδοποιήσει ότι αποκλείεται ε, να ε, μπει σε λεπτομέρειες για την νομοθεσία. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε για τους άλλους ομιλητές. Δηλαδή δεν έχετε καμία ερώτηση για οποιονδήποτε άλλον. Εάν όχι, α, παρακαλώ. Και να μας πείτε και ποιος είστε. Γεια σα, η Σέντε ε, είμαστε από τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ε, Κολομβία. Απευθύνομαι στον κύριο Σέρχιο Κολονάντο. Έγιναν πολλέ απεργίε στην Κολομβία, στην εξορρυκτική βιομηχανία πρόσφατα και μπορείτε, αν έχετε την καλοσύνη, να μα εξηγήσετε γιατί έγιναν όλε αυτές οι απεργίε και ποια ήταν ε, η αντίδραση της Κολομβίας, της κυβέρνηση και της Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Sí, recientemente el gobierno colombiano expidió un... Μάλιστα, πρόσφατα η, η κολομβιανή κυβέρνηση πέρασε ένα νομοσχέδιο με στόχο να ε, αναχαιτήσει την παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα ε, να ε, σταμα... διακόψει τη λειτουργία μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε η βιομηχανία στην αρχή μπορεί ε, να φάνηκε ως μια θετική δράση όμως ε, ήταν ισχυρότατες ε, οι αντιδράσεις όχι μόνο από τους ιδιοκτήτες των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων αλλά και αντίδραση όλων όσων ζουν από αυτό. Το πάλο μινέρο το περίφημο, δηλαδή η ε, ανάσχεση εργασίας, ε, οι απεργίες ε, που έγιναν, ε, οδήγησαν μετά από πολλές διαπραγματεύσεις σε μία συμφωνία ε, ως προς αυτά τα κατασταλτικά μέτρα της κυβέρνησης της Κολομβίας. Ο στόχος είναι καλή η πρόθεση, έτσι είναι ο έλεγχος ε, της παράνομης δραστηριότητας. Το πρόβλημα όμως ε, είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κοινωνικό ε, πλαίσιο, διότι οι σειράξει αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο στην Κολομβία και πρέπει να συνυπολογίζεται. Ε, πρόεδρος, εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο επίγον ερώτημα, θα ζητήσω από τη ΣΑΣΚΕ και από τον Τέτε να μοιραστούμε και μαζί μας κάποιες σκέψεις μετά και από την παρέμβαση του Επιτρόπου De Huchtum, ώστε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες του πρώτου πάνελ ή να μας πούν όλα αυτά που θέλανε να πούνε, αλλά δεν τους εδόθη η ευκαιρία λόγω έλλειψης χρόνου. Σας και θα ακούσουμε ένα πρώτο και στη συνέχεια τον τέτε. Δύο είναι οι παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Και ο Τέτε και πώς λένε, ξέχασα τον όνομα, ο Σέργιο. Ξεκαθάρισαν ότι για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη ε, πρέπει να παραχθεί εισόδημα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης από την εξορρυκτική βιομηχανία. Μόνο έτσι μπορούν να υποφεληθούν οι χώρες από αυτή τη δραστηριότητα. Μόνο έτσι θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και έτσι εφαρμόστηκε η νομοθεσία για το περιβάλλον ε, και για την έγκαιρη προειδοποίηση. Όταν βλέπουμε τώρα για το μηχανισμό διεξαγωγής ελέγχων, ε, ξέρουμε ότι δεν επαρκεί για να ε, ρυθμίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ ευρύτερα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εξετάζει την εμπορική, την επενδυτική πολιτική της, την κανονιστική πολιτική της ε, για αυτό τον κλάδο, για να εξετάσει ποιες αυτές τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τώρα, για το σύστημα υποχρέωσης ελέγχου θα μπορούσα να σας πω θα συμπληρώσει βέβαια και ο ΤΕΤΕ κάποια πράγματα. Τι θα θέλαμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών για να μεριμνήσει ούτω ώστε τα ωφέλη να τα καρπώνονται αυτέ οι χώρε ε, και να μην υπάρχει η εξόριξη φυσικών πόρων τη χώρα χωρί κανένα όφελο για αυτήν. Ε, ξέρω ότι το είπα και νωρίτερα, το 2001... Ε, ο Όμιλος ε, Παγκόσμιας Τράπεζας ζήτησε την αναθεώρηση, μια διετή αναθεώρηση της κατάστασης. Έγιναν πάρα πολλές διαβουλεύσεις, επιτόπου επισκέψεις και... Ε, περιβαλλοντικές ε, ΜΚΟ, μικρών ε, κοινωνικές ΜΚΟ, μικρών οργανώσεις από τον τομέα της διακυβέρνησης, εκπρόσωποι των εταιριών μετήχαν σε αυτήν την έρευνα σε σχέση με τους απότερους στόχους. Να σας διαβάσω ποιοι είναι αυτοί οι απότεροι στόχοι, γιατί πιστεύω ότι και εμείς πρέπει να τους έχουμε κατά νου όταν εξετάζουμε το μέλλον της εξορρεκτικής βιομηχανίας εδώ στην Ευρώπη, εξετάζω τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, να το, στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, ε, κρατέα εταιρική σχέση ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση. Πρώτο στόχο. Δεύτερον, να υπάρξει μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ούτω ώστε να υπάρξει μια αντιστάθμιση των οικονομικών στόχων, ε, ταυτόχρονα ανακούφιση από τη φτώχεια και τρίτον, ε, ε, η πνευματική στόχη της ζωής κατά τη διαστολή με τους οικονομικούς στόχους που μπορεί να έχουμε. Αυτή είναι η τριστόχη και εγώ ανησύχησα κατά τι όταν είπε ο Επίτροπο ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και να βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη. Εντάξει, αληθεύει αυτό σε ένα κάποιο βαθμό. Δείτε όμω ε, τον εμφύλιο πόλεμο που γίνεται στην Κεντρική Αφρική. Ωραία, ποιο είναι το εφαλτήριό μα. Ε, το ίδιο. Αν δούμε το Κόγκο, ποια πραγματικότητα χρησιμοποιείτε εσεί ω εφαλτήριο ακριβώ, διότι αυτέ οι χώρε ε, εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Οι άνθρωποι εργάζονται με κίνδυνο τη ζωή του, ώστε να γίνονται σεβαστοί τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να του ακούμε. Λοιπόν, να σα πω ποια είναι η πραγματικότητα, ότι δεν εισακούονται προ το παρόν και είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία που έτσι περαιτέρω υπονομεύει την κοινωνία αντί να την υποστηρίζει. Ε, δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε εσά και λέει Πρόεδρος. Ε, τέτε είσαι εκεί μόνος σου στην Κάνα, σε, αυτή την, σε αυτό το άδειο δωμάτιο, άκουσες ε, φαντάζομαι τον Επίτροπο Τεχούχτ ε, και τους ε, συναδέλφους. Δύο λεπτάκια αν θα μπορούσες να μοιραστείς τις σκέψεις σου μαζί μας. Um, just two quick points uh, to, to say. The first thing is to return to the commissioners of the vision that whatever they, they want to do in relation to conflict uh, has to be balanced with the You have to repeat the last sentence. Have Τέτε, πρέπει να επαναλαβείς τις ε, ε, τελευταίες ε, προτάσεις γιατί χάθηκε ο ήχος.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 Εκτιμούμε την παρουσία σας. Ε, την παρουσία σας. Θα αλλάξουμε εδώ τώρα θέσεις ε, στο βήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ένα χειροκρότημα γιατί μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. I'll invite... I'll invite... Θα καλέσω τώρα την ε, κυρία Αν Φρανσουάζ Μελό, ε, η οποία είναι επικεφαλής ε, της Unit F3, καθώς επίσης και τον Ρομπέρτο Ριντόλφι, ο οποίος είναι διευθυντής του τμήματος για την αηφόρα ανάπτυξη και την ανάπτυξη στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Τώρα, εάν εσείς θέλετε να μείνετε κάπου γιατί την παρουσίασή σας πρέπει να την κάνετε ε, από τη θέση σας, ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα προχωρήσουμε με ταχύτητα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ καλό κορίτσι, λέει η Πρόεδρος, και πάντα σέβομαι τα χρονικά περιθώρια. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει σε 25 λεπτά από τώρα. Η κυρία Αν Φρανσουά Μελό δεν μας κρύβεται, αλλά είναι εκεί πίσω με τον υπολογιστή της. Και θα δείτε, θα κάνει μια παρουσίαση PowerPoint. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή πλέον. Ε, ε, δυστυχώς έκανα λάθος υπολογισμό του χρόνου, αλλά τώρα δεν θα ε, μπορώ να σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ την ε, τους εισηγητές ε, για τα θέματα τα οποία έθιξαν σήμερα το πρωί με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ε, και με στόχο βεβαίως να υπάρξουν πιο καλές εμπορικές πρακτικές και να δείχνουν και οι εταιρείε μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο νέες υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείε. Η πρώτη είναι αυτό το σύστημα του counter reporting ε, δηλαδή η αναφορά αναχώρα, country by country reporting, Πρόκειται για ένα κεφάλαιο της ε, νέας λογιστικής ε, οδηγίας, την οποία θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Το κείμενο άλλωστε έχει εγκριθεί. Και η δεύτερη υποχρέωση αναφέρεται πάντα στις προτάσεις ε, της ε, Επιτροπής. Πρόκειται για ένα ε, κείμενο το οποίο συζητιέται και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις, στην αναφορά των non-financial information από τις πληροφορίες, δηλαδή μη χρηματοδοτικού χαρακτήρα από τις εταιρείες. Ποιος είναι ο στόχος μας ε, ε, όταν θέλουμε αναφορά αναχώρα, country by country reporting. Θέλουμε να γίνουν ε, οι εταιρείες αλλά και οι χώρες, οι κυβερνήσεις οι οποίες ε, εκμεταλλεύονται τους ε, φυσικούς ε, πόρους να γίνουν, λέω, πιο υπεύθυνες, έτσι ώστε οι ντόπιε κοινότητες να έχουν γνώση του τι συμβαίνει και επίσης να γνωρίζουν και οι κάτοικοι και οι αυτόχθονες τι πληρώνουν οι εταιρείες και ποιο είναι τελικά το τίμημα το οποίο καταβάλλεται και εάν ε, ε, πληρώνουν ένα σωστό τίμημα για την εκμετάλλευση την οποία έχουν. Εάν δηλαδή εκμεταλλευόμενοι τους ε, φυσικούς τους πόρους, τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν στο δικό τους έδαφος, καταβάλουν ένα δίκαιο σωστό αντίτιμο. Με ποιο τρόπο ελπίζουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αυτή η νέα υποχρέωση της λογιστικής οδηγίας αναφέρεται στις μεγάλες εταιρείες, τις οποίες, ε, ε, στις οποίες ε, πλέον δίνουν κάποιες υποχρεώσεις. Όταν λέμε μεγάλες εταιρείες, αναφερόμαστε σε εταιρείες οι οποίες έχουν πάνω από 250 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών πάνω από 100.000 ευρώ. Ε, μπορεί να είναι ε, ντόπιε εταιρείε ή μπορεί να είναι ε, εταιρείε ευρωπαϊκέ ή εταιρείε οι οποίε βρίσκονται σε τρίτε χώρε. Πρόκειται για εταιρείε οι οποίε βεβαίω έχουν σαν, κύριο, σαν κύρια ενασχόληση την εκμετάλλευση των δασών, ε, πετρελαιοπηγών και εξορρυκτικής ε, διαδικασίας. Ε, αυτό το, το, στοιχείο των, ε, ε, της ξυλίας μας διαφοροποιεί και από την αμερικανική πράξη την Dodd Frank. Αυτές οι εταιρείε λοιπόν θα υποβάλουν ε, πλέον μια ξεχωριστή έκθεση η οποία θα αναφέρεται στο τίμημα το οποίο καταβάλουν στις χώρες με τις οποίες ε, συνεργάζονται και με τις οποίες έχουν συμβάσεις. Αναφερόμαστε σε πληρωμές οι οποίες ξεπερνούν τις 100.000 ε, ευρώ σε είδος ή σε χρήμα. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους και βεβαίως ζητούμε από τις ε, κυβερνήσεις να μας δώσουν ε, συγκεκριμένες πληροφορίες ανά project Έγινε πολλή συζήτηση για, την, ε, για τον ορισμό αυτό ε, και καταλήξαμε στο ότι ε, ως project θεωρείται οποιαδήποτε είδους δραστηριότητα. Και όταν αναφερόμαστε σε πληρωμές, βεβαίως αναφερόμαστε στους τίτλους παραγωγής, στους φόρους και τα μισθώματα, στα μερίσματα, άδειες εκμετάλλευσης κτλ. Όπως ε, είπα και προηγουμένως, ε, οι Ηνωμένε ε, Πολιτείες έχουν ήδη νομοθεσία Πρόκειται για το τμήμα 1504 της Dodd-Frank Act. Και σήμερα, αυτό το καλοκαίρι υπήρξε και μία δικαστική απόφαση ε, σχετικά με εσφαλμένη ερμηνεία της Dodd-Frank ε, Act όσον αφορά την δημοσιοποίηση ε, όλων αυτών των λεπτομεριών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επιθυμούν μονάχα η SEC να έχει αυτές τις πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ζητούμε πάντα δημόσια πληροφόρηση, αλλά βεβαίως ε, θα γίνει μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τις ε, ρήτρε ε, ομοτιμίας, γιατί πρόκειται εδώ για δυνατότητα που δίνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες να προσαρμοστούν στις και οι οποίες θεωρούνται ομότιμες εταιρείες να μην χρειάζεται να περάσουν από τον ε, συγκεκριμένο ε, έλεγχο και επομένως αυτή η ρήτρα ισοτιμίας είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης ε, σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι υπήρχε ήδη η λεγόμενη Extractive Industries Transparency Initiative, η πρωτοβουλία διαφάνειας δηλαδή ε, για τις εξορρυκτικές ε, βιομηχανίες, η ITI, βάσει της οποίας όλες οι εταιρείε οι οποίες δραστηριοποιούν το επιτόπου ήταν υποχρεωμένες να δώσουν κάποιες πληροφορίες, ε, αλλά οι αμφιτρίωνες χώρες δεν είχαν την υποχρέωση να συνυπογράψουν αυτήν την έκθεση. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα, πού βρισκόμαστε. Αυτή η υποχρέωση αναφοράς όπως σας είπα και προηγουμένως, αναφέρεται ε, στην ε, λογιστική οδηγία. Έχουν είχαν ένα χρόνο οι χώρες για την ενσωμάτωση στην νομοθεσία τους, Ιούλιος δηλαδή 2013, ε, μέχρι τον Ιούλιο του 2015 θα πρέπει όλες οι χώρες μέλη να έχουν ενσωματώσει την ε, νομοθεσία το 2016 θα έχουμε την πρώτη ενδεχόμενη εφαρμογή και το 2018 ενδεχομένως αναθεώρηση του συστήματος. Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε μονάχα στις εταιρείες οι οποίες ήδη ε, είναι ενεργές και δραστηριοποιούνται ε, στην εξόριξη. Ε, σιγά σιγά όμως θα υπάρξει διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής με τις ε, κατασκευαστικές εταιρείες ε, και άλλες. Ε, θα δούμε, θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα πού βρισκόμαστε και ποια είναι, ποιος είναι και ο συσχετισμός με το αμερικανικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει και τις συζητήσεις για το non-financial reporting. Ήδη υπάρχει ένα κεφάλαιο στην οδηγία που ανέφερα προηγουμένως αλλά ε, δεν έχει πάρει τελική μορφή. 10% των μεγάλων ε, ε, εταιριών τούτη τη στιγμή ήδη κάνουν, δημοσιεύουν εκθέσεις οι οποίες δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο, αναφέρονται στο περιβάλλον, στην, στα κοινωνικά μέτρα κτλ. Υπάρχουν επίσης χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, η Δανία, η Ισπανία όπου η νομοθεσία είναι και πιο δεσμευτική όσον αφορά ε, αυτήν την ε, δυνατότητα αναφοράς. Εμείς θέλουμε να τροποποιήσουμε την νομοθεσία έτσι ώστε να υποχρεωθούν όλες οι μεγάλες εταιρείες να έχουν διαφάνεια όσον αφορά ε, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα ζητήσουμε λοιπόν να ε, δώσουν στοιχεία όσον αφορά τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει, τους κινδύνους που συνδέονται με τις ε, ε, πολιτικές αυτές και αναφέρονται πέντε συγκεκριμένα πεδία, το περιβάλλον, κοινωνικά ζητήματα και οτιδήποτε σχετίζεται με το προσωπικό, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και τέλος διαφοροποίηση όσον αφορά την ε, σύνθεση ε, των διοικητικών συμβουλίων. Δεν αναφερόμαστε μονάχα στην ίση εκπροσώπηση ανδρών γυναικών αλλά και ίση εθνοτική εκπροσώπηση κτλ δεν υποχρεώνουμε τις εταιρείες να κάνουν συγκεκριμένη, να εφαρμόσουν συγκεκριμένη πολιτική, απλώς υποχρεώνουμε τις εταιρείες να δουν την πολιτική τους ε, με μεγαλύτερη ε, υπευθυνότητα. Βεβαίως, βεβαίως μας ενδιαφέρει να μην αυξήσουμε υπερβολικά το διοικητικό άχθος των εταιριών, κυρίως ε, στα πλαίσια ε, αυτών των χαλεπών καιρών, της κρίσης που ε, διανύουν οι χώρες. Λέμε λοιπόν ότι μονάχα οι πολύ μεγάλες εταιρείες θα οφείλουν, ε, θα έχουν αυτή την ε, υποχρέωση. Ε, αναφερόμαστε σε 18.000 περίπου εταιρείε οι οποίες έχουν πάνω από 500 εργαζόμενους, εταιρείε οι οποίες είναι εγκατεστημένε στην Ευρώπη, αλλά και ξένες εταιρείε οι οποίες όμως έχουν παρουσία ε, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μία συσχέτιση και με την οδηγία για την ε, διαφάνεια που αναφέρεται στις εισηγμένες εταιρείες. Τώρα, εάν ε, οι εταιρείε οι οποίες, εάν ε, οι θεωρούν ότι δεν έχουν ή δεν επιθυμούν να έχουν συγκεκριμένη πολιτική στον ένα ή στον άλλο τομέα, στο ένα ή στο άλλο πεδίο ε, στο οποίο εμείς ζητούμε να γίνεται αναφορά, τότε έχουν τη δυνατότητα να μην υποβάλουν έκθεση για το θέμα αυτό. Δεν ζητάμε άλλωστε τεράστιες εκθέσεις, ζητάμε να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τις πολιτικές πρακτικές που εφαρμόζονται, την εκτίμηση των κινδύνων, τους κινδύνους που συνδέονται με τις οποιασδήποτε πολιτικές, τα αποτελέσματα κτλ. Οι εταιρείε έχουν την ε, δυνατότητα, έχουν την ελευθερία να βασίσουν την έκθεσή τους σε εθνικά ε, στοιχεία, σε εθνικές αρχές ή διεθνή πρότυπα όπως ας πούμε το Global Reporting Initiative ή ε, το, το σύστημα αναφοράς ε, το, του ΟΣΑ κτλ. Λοιπόν, όπως ε, ε, σας είπα φέτος, τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει η πρόταση αυτής της ε, οδηγίας. Ε, θα υπάρξει συζήτηση και στο Συμβούλιο και παντού ε, και ε, θα έχουμε μάλλον την πρώτη εφαρμογή από τις εταιρείες το 2015 με την προϋπόθεση ότι θα τεθεί θα, σε ισχύ το 2014. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βέβαια ήταν πολύ καλό που ακούσαμε μερικά για το, τι, για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μετά την ε, απόφαση που πήραμε το καλοκαίρι, την ψηφοφορία που έγινε για την οδηγία και πώς εφαρμόζεται αυτή. Μετά από 10 χρόνια ε, στον τομέα αυτό μερικά πράγματα συνεχίζουν να με εκπλήσουν. Τώρα προχωρώ στο Ρομπέρτο Ριντόλφι, είναι διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Έχει ασχοληθεί με πολλά θέματα από αυτά που μας απασχολούν και μας και ε, την Επιτροπή μας. Είστε ο τελευταίος ομιλητής μας κύριε Ριντόλφη και δεν φταίτε εσείς βέβαια αλλά δεν έχετε και πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί ευρωβουλευτές κυρίες και κύριοι χαίρομαι που παίρνω μέλος σε αυτή την ακρόαση ε, γιατί για μένα αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή χτες ε, ανέλαβα ως διευθυντής ε, στη EuroPaid για την βιώσιμη ανάπτυξη και, μπορώ, και πήγα και στη Ιουγκάντα και μπορώ να σας πω αρκετά πράγματα από εκεί. Ξεκινάμε σαν από την βασική ιδέα ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα είναι η κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη. Αν δεν το πιστέψουμε αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο ιδιαίτερος, ο ιδιωτικός τομέας με τον οποίο θέλουμε να συνεργαστούμε. Αυτό περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της, που ενέκρινε και το Συμβούλιο και που ονομάζεται ε, Agenda for Change και εμείς τώρα καλούμε θα, σαν Κομισιό να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά πρέπει να κάνουμε, δύο, να κάνουμε αγώνες σε δύο μέτωπα. Πρώτα πρώτα πρέπει να κάνουμε ε, κάποια πράγματα για να δημιουργήσουμε ένα καλό περιβάλλον και μια καλύτερη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία να μπορεί να δράσει ο ιδιωτικό τομέα. Και δεύτερον θα πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους σύνδεσης και σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Ε, ε, ε, ξέρουμε ότι ενώ η Ευρώπη περνάει μια εποχή κρίσης υπάρχουν άλλες περιοχές ε, του πλανήτη στην Αφρική λόγου που ε, έχουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης μόνο που η ανάπτυξη είναι μόνο στα νούμερα για το κεφάλαιο αν θέλετε και δεν δημιουργούν νέες θέσεις δεν δημιουργεί νέες θέσεις γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και το τι θα κάνουμε εμείς και πόσο ευρώ ο ιδιωτικός βοηθήσει και πώς θα διατηρήσουμε μια τεράστια μια διαφάνεια για να πείσουμε και τις εταιρείε σχετικά η διαφθορά που Δυστυχώς ε, είναι κάτι το οποίο συζητείται πολύ στις επαφές μας στο, με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διαφθορά είναι... Ε, χρειάζεται δύο άτομα και αυτός που διαφθείρεται και υπάρχει αυτός που διαφθείρεται και αυτός που διαφθείρει λοιπόν να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας Πρέπει, να δράσουμε επίση στο τομέα των προτύπων. Θέλουμε να παρθούν αποφάσεις για τα πρότυπα ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε δίκαιο θεμητό εμπόριο. Fair trade. Θέλουμε λοιπόν να... Ε, επίσης υπάρχει όπως ξέρετε η ε, ε, Εμπόριο εταιρική ευθύνη, ε, κοινωνική ευθύνη την οποία προωθούμε στην Ευρώπη ιδιαίτερα πιστεύουμε ότι πρέπει να οριστούν σχετικά πρότυπα η Γενική Διεύθυνση Μάρκτα ασχολείται με αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε υποχρεωτικές ε, τις, ε, ε την κοινωνική ευθύνη μέχρι στιγμής όλα είναι προαιρετικά στον τομέα αυτό αλλά ε, ίσως πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω να μην κοροϊδευόμαστε όλα στη Αφρική και αναφέρομαι σε αυτή γιατί είναι η Ήπειρος που γνωρίζω καλύτερα ε, η, η, Ευρώπη ε, πιέζει στην Αφρική ας πούμε για θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αλλά βλέπουμε ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν το ίδιο γίνεται με την κοινωνική ευθύνη και ε, πολλές φορές ε, βλέπουμε εταιρείε του ιδιωτικού τομέα που αρνούνται να ακολουθήσουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές αλλά στην πραγματικότητα αλλά και βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είμαστε και ο μόνος παίκτη. Για τα θέματα αυτά δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Υπάρχουν και άλλοι. Προσπαθούμε να προχωρήσει η ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας αυτή η decent work agenda που έχουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη ε, αν θέλετε μεγαλύτερο σεβασμός προς τον εργαζόμενο καλύτερα εργασιακά στάνταρτ πρότυπα παραδείγματος χάρη. Προσπαθούμε να τα βάλουμε αυτά σε όλα τα προγράμματα συνεργασίας. Προσπαθούμε αυτά τα να βάλουμε δράση στα προγράμματά μας για να προωθήσουμε υπεύθυνα προγράμματα. Παράδειγμα, υπάρχει το πρόγραμμα Switch Asia για την Ασία, για την περιοχή της Ασίας που τώρα εξ, διευρύνεται και προς την Μεσόγειο και προς προς κάποιες περιφέρειες της Αφρικής το οποίο είναι άξιο να το παρακολουθήσει κανείς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνοδεύσουμε τις ε, ε, εθνικές προσπάθειες που κάνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύουμε ότι πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να προχωρούμε. Αλλά ποια κοινωνία των πολιτών, όχι της Ευρώπης, της χώρας στην οποία δουλεύουμε, διότι αυτοί ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να ε, προωθήσουμε τις ιδέες αυτές. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ε, είναι υπεύθυνη για το διεθνές πλαίσιο και για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις <coughs> και εμείς προσπαθούμε να ε, δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ε, κοιτάξτε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι οι δημόσιες προμήθειες και οι σχετικοί διαγωνισμοί που γίνονται και τα λοιπά. Τα περισσότερα κράτη ε, προβαίνουν στη διαδικασία αυτή και εξαρτώνται όλο και λιγότερο από τη βοήθεια. Γι' αυτό η βοήθεια δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολιτικοί εταίροι των χωρών αυτών, είμαστε αναπτυξιακοί εταίροι. Δεν είμαστε απαραίτητο χορηγοί, δωρητές, donors όπως άλλοι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά η εξορρυκτική βιομηχανία. Και θα ήθελα κυρία Πρόεδρε για να μην χάνω το χρόνο σας να σας πω να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό ε, κυρία Πρόεδρε. Είναι θέμα των κυβερνήσεων, των, των, της κοινωνίας των πολιτών των χωρών αυτών ε, ε, να προχωρήσουν. Ε, δεν πρέπει οι χώρες αυτές να φροντίσουν για να μην, από, να μην καταλήξει κατάρα η ύπαρξη φυσικού πλούτου σε αυτές τις χώρες. Το παράδειγμα της Ιουγκάντα είναι πολύ σημαντικό ε, ε, όπου δεν ε, καταφέρνουμε πολλά να κάνουμε και να πούμε. Υποστηρίζουμε τη διαδικασία ε, για το που βοήθησε στο, στον τομέα των διαμαντιών έχουμε Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και η παρουσίαση εκθέσεων και συγκεκριτικών εκθέσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών είναι πολύ σημαντικά. Η διαφθορά είναι ε, μεγάλο θέμα και βάσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η διαφάνεια είναι ε, που ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βεβαίω αυτά όλα συνδέονται με την ασφάλεια, διότι στην Κεντρική Αφρική δίχως ασφάλεια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάντως η προσέγγιση την οποία υιοθετούμε τώρα για την ε, ανάπτυξη ε, ε, έχει και κάποιους περιορισμούς βεβαίως που σχετίζονται και με τα εισοδήματα των διαφόρων χωρών από το, το πετρέλαιο και τα φυσικό αέριο τα εισοδήματα των χωρών της Αφρικής θα αυξηθούν σημαντικά θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και να τα έχουμε υπόψη μας αυτά όλα όταν συζητούμε με τις χώρες αυτές ε, σε όλα τα επίπεδα και σε σχέση με τον δημόσιο τομέα και σε σχέση με τον ιδιωτικό ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι εύκολη η δουλειά μας. Εμείς σαν Κομισιόν θα για το ρόλο του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη. Θα κάνουμε μια ανακοίνωση του χρόνου και προσπαθούμε να ε, προωθήσουμε και την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ολοκληρώνουμε. Δεν είναι δυνατόν σε δυόμιση ώρες να λύσουμε ή να κάνουμε το γύρο όλων αυτών των σημαντικών θεμάτων. Και ξέρω ότι θα με μισήσετε γιατί δεν δίνω τη δυνατότητα ε, σε άλλους να μιλήσουν ή να υποβάλουν ερωτήματα. Αλλά να μην λησμονούμε ότι έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας όχι, όχι, δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε κανέναν. Λοιπόν, ε, στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά άρθρα, ε, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα χαράξουμε με τουάζου στο χέρι μας, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχει η ο κανόνας, το άρθρο που λέει ότι ο κανόνας για την ανάπτυξη είναι η εκρίζωση της φτώχειας και έχουμε και το άρθρο 208 που λέει ότι όλες ε, οι ε, δραστηριότητες δεν μπορούν ε, να, οποιαδήποτε δραστηριότητα δηλαδή, δεν μπορεί να αντιταχθεί σε αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο της εκρίζωσης της ένδυας. Έχουμε λοιπόν το νομοθετικό πλωστάσιο το οποίο είναι στο πλευρό μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και το ακούσαμε σήμερα ότι αυτό σου ανοίγει το δρόμο ε, για ελεύθερη ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ε, Ακούσαμε προηγουμένως ε, το θέμα των προσφύγων που δεν μένουν στο Μαλί ή δεν μένουν ε, στην Γκάνα και ο κύριος ε, Ρεντόντο Δελγάδο έκανε την ίδια παρατήρηση επίσης και ο μιλητής που μόλις ακούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, εάν έχουμε μια σωστή αναπτυξιακή προώθηση, τότε μονάχα θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Εγώ εκπονώ έκθεση με τον ίδιο τίτλο. Πρόκειται για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο με την ακρόαση. Επομένως, Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, ε, να μου το στείλετε ε, με mail, να μου το δώσετε γραπτά, έτσι ώστε να μπορέσω ε, τον προβληματισμό σας να τον βάλω και στην έκθεσή μου. και ίσως αν ε, ε, εκπονηθεί η έκθεση μέχρι τον Δεκέμβριο να συμπέσει και με την ε, ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ο Επίτροπος Ντεγούχτ. Τελειώσαμε εδώ. Ελπίζω ότι θα έχω ανάδραση από την πλευρά σας, ότι θα μου στείλετε όλα τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ βεβαίως πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ και τους οργανωτές.